Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ορίσατε. Συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση, αλλά όπως γνωρίζετε παρακολουθούμε τις εκλογές στην Ουκρανία σε τρεις εβδομάδες και τα ουκρανικά μέσα μαζικής ενομέρισης θα ήθελα να γνωρίζουν ε, πώς και πότε θα παρακολουθήσουμε τις ε, τοπικές εκλογές για πρώτη φορά μετά την Γεωργία. Όπως μπορείτε να δείτε στην ημερήσια διάταξη ε, σήμερα επικεντρωνόμαστε σε δύο ζητήματα. Ο ένας είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των Ηνωμένων Εθνών, πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερα τους στόχους εξωτερικής πολιτικής μας και Έχουμε και ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, το οποίο έχει αλλάξει λίγο. Η ανταλλαγή απόψεων με τον Κριστιαν Λέφνερ για τις ε, σχέσεις για την Κούβα. Ποιος είναι υπεύθυνο για τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κούβας το θέμα σχετικά με την επιστημονική διπλωματία έχει αναβληθεί για κάποια άλλη συνεδρίαση. Θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν απευθεία στο σημείο 3 που είναι η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έξεσης που έχει ε, καταρτήσει ο συνάδελφος Παύο Βαϊράινεν. Ε, αρκετοί συνάδελφοι έχουν εργαστεί αρκετά ε, σκληρά τους προηγούμενους μήνες. Πρόκειται για μια σημαντική έκθεση που προσπαθεί να δει πώς μπορεί να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο καλύτερα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της επίτευξης των κυρίων στόχων ε, εξωτερικής πολιτικής μας. Έχουμε 322 τροπολογίες, ε, πέντε επιτροπές γνωμοδότησαν επί της έκθεσης αυτής και γνωρίζουμε ότι ο εισηγητής και η σκιώδης ε, υπέβαλαν 24 συμβαστικές τροπολογίες για την έκθεση αυτή. Ε, επιπλέον θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων η έκθεση αυτή ε, επισημάνθηκε ότι δεν αποτελεί την επίσημη υποβολή της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά πρόκειται για μια εξέταση για να δούμε πώς μπορούμε το σύστημα αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως καταλήτη και να μεγιστοποιήσουμε ε, την επιρροή μας στα Ηνωμένα Έθνη ε, που είναι παγκόσμιος οργανισμός αλλά και στον παγκόσμιο προσκήνιο εν γέννη. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον κύριο Βαϊράινα να μας κάνει μια παρουσίαση του τι ακριβώς συνέβη εν μεταξύ και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω επίσης ότι αύριο το πρωί θα ψηφιστεί η έκθεση. Κύριε Βαϊράινα να έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ε, εισαγωγή για την, το σκεπτικό της έκθεσης. Δεν πρόκειται για τη μετήσια έκθεση για τα Ηνωμένα Έθνη, πρόκειται για μια έκθεση η οποία στόχο έχει να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις δυνατότητες που διαθέτει να επηρεάσει τις διεθνείς εξελίξεις στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Αρχικώ είχα προτείνει να είναι ευρύτερο ο τίτλο τη έκθεση ε, και να λαμβάνει υπόψη του και τον παγκόσμιο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατόπιν όμω περιοριστήκαμε στα Ηνωμένα Έθνη Διαγωνός που στην πραγματικότητα δεν περιόρισε πάρα πολύ ε, την έκθεση, γιατί το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών καλύπτει όλες τις τη της ε, πολύπλευρης συνεργασίας. Αυτό το οποίο εκκρεμεί τώρα είναι οι διμερείς μας σχέσεις με ε, χώρες και ομάδες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτυχή όμως των παγκοσμίων ε, πολυμερών θεμάτων καλύπτεται εδώ στην έκθεση αυτή. Προκειμένου λοιπόν να ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας για την επίτευξη των στόχων μας από πλευράς εξωτερικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει καταρχάς να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των Ηνωμένων Εθνών και του συστήματός τους. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα για παγκόσμια διακυβέρνηση να ενισχυθούν ε, τα Ηνωμένα Έθνη στο παγκόσμιο πλαίσιο. Και επίσης θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αυξήσουμε και την επιρροή μας ε, στο ε, σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό προσπαθεί να προτείνει η έκθεση. Η δομή της έκθεσης είναι πολύ απλή. Πρώτα ανέφερα τους στόχους πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στη συνθήκη. Μετά υπάρχει μια ε, γενική περιγραφή του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και μετά μια παράγραφος που αναφέρεται στο ε, πώς μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι της έκθεσης αυτής. Το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών έχει δύο πυλώνες από τότε που ε, ε, διατυπώθηκε η χάρτα πριν από 70 ε, χρόνια. Έχουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας και το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης κάνω κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το Συμβούλιο Ασφαλείας και να βελτιώσουμε τη λειτουργία του. Αλλά βεβαίως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εκβάθρον αλλαγή του Συμβουλίου Ασφαλείας ε, στην πράξη θα είναι αδύνατον να γίνει. Αυτό ε, που προτείνουμε είναι τι θα μπορούσε να γίνει στις παρούσες συνθήκες. Κατόπιν γίνονται κάποιες προτάσεις για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την οικονομική και κοινωνική πτυχή του συστήματος των ΗΕ. Στην έκθεση ε, είχα αρκετά φιλόδοξες ιδέες θα ήθελα να σταθώ σε τρεις εξ αυτών. Καταρχάς ε, προτείνω να υπάρχει και ένα κοινοβούλιο των Ηνωμένων Εθνών το οποίο θα λαμβάνει αποφάσεις και το οποίο μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να γίνει ένα παγκόσμιο κοινοβούλιο. Δεν υπήρξε βέβαια υποστήριξη από την πλειοψηφία στις διαπραγματεύσεις ούτε καν αυτή η ιδέα της ε, κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Ο κύριος Γιολάινεν ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δύο φορές έχει δεχτεί την ιδέα μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης, αλλά αυτή τη φορά τουλάχιστον στις διαπραγματεύσεις με τους κοιόδης ηγητές δεν είχα υποστήριξη της πλειοψηφίας. Θα ψηφιστεί βέβαια ε, υπάρχει ξεχωριστή ψηφοφορία, δεν περιλαμβάνεται στις συμβαστικές τροπολογίες η πρόταση αυτή. Η δεύτερη φιλόδοξη ιδέα μου ήταν να υπάρξει ένα οικονομικό και κοινωνικό συμβούλιο το οποίο θα γίνει ένα συμβούλιο βιώσιμης ανάπτυξης το οποίο θα καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες πτυχές συνεργασίας εκτός της ασφάλειας και προτείνω αυτό το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης να έχει την ίδια δομή και το ίδιο στάτους με το Συμβούλιο Ασφαλείας. Να υπάρχουν μόνιμα μέλη ε, που θα είναι οι μεγάλες οικονομικές δυνάμεις ε, στον κόσμο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να υπάρχουν και περιτροπής μέλη. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα μπορεί να έχει μια πολύ ισχυρή επιρροή στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό υπ' αυτή τη μορφή, αλλά στην παράγραφο 5, στη συμβιβαστική τροπολογία 8, καταλήξαμε σε μία μάλλον ικανοποιητική διατύπωση και έτσι αναφέρεται ότι το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο θα πρέπει να ενισχυθεί και αυτό θα πρέπει να γίνει καταρχάς μέσω διαρθρωτικών και λειτουργικών μεταρρυθμίσεων των, ε, του βασικού οργάνου που είναι αρμόδιο για αυτό το, ε, τα καθήκοντα, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, δηλαδή να γίνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, χωρίς να αναφέρουμε ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και κατόπιν στην επόμενη φράση Καλούνται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενίσχυση του ρόλου του στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο μετατρέποντάς το σε ένα Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αναφέρεται δηλαδή η αλλαγή του ονόματος ε, του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου. Αυτό είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο συμβαστικό κείμενο. Δεν είναι αυτό το οποίο επιθυμούσα, αλλά είναι πολύ κοντά. Επομένως θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε αυτή την ιδέα στο μέλλον. Κατόπιν, η τρίτη μου φιλοδοξία κατά την εκπόνηση αυτού του κειμένου ήταν να οργανώσουμε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λίγο καλύτερα όσον αφορά τα παγκόσμια ζητήματα. Σε αυτό το σχέδιο έκθεσης, ε, το έχουμε μάλιστα και στις συμβασικές τροπολογίες, καταρχάς επικροτούμε την οργάνωση αυτή σε θεματικέ ονότητε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε κλάστερ. Έτσι ε, υπάρχουν επίτροποι που είναι αρμόδιοι ε, για να καθορίσουν όλες τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μαζί με όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και εδώ τονίζουμε ότι οι πολιτικές με παγκόσμια διάσταση θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών τη συγκεκριμένη αυτή θεματική ονότητα. Και μετά, στη συμβαστική τροπολογία 16, καλούμε την ύπατη εκπρόσωπο να συμπεριλάβει στην ετήσια έκθεσή τη ε, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και την ε, Πολιτική Ασφάλεια και Άμυνα να υπάρχει ειδική μνήμα για την παγκόσμια διάθεση των πολιτικών μα. Και μετά, στην επόμενη παράγραφο, αναφέρουμε ότι είμαστε τη άποψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τι παγκόσμιε προκλήσει τον ίδιο συνολικό τρόπο όπως ε, οργανώνει ε, τις εργασίες της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να οργανώσει και αυτό τις εργασίες του καταλήλως. Ενθαρρύνει όλες τις επιτροπές που έχουν εντολή που καλύπτει και εξωτερικές πολιτικές ε, και παγκόσμια διάσταση να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη τομέα της έκθεσης της υπάτης εκπροσώπου που είναι αρμόδια για την έκθεση αυτή. Δηλαδή η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων βάσει αυτής της διατύπωσης θα συντονίζει το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ζητά από όλες τις αρμόδιες επιτροπές να γνωμοδοτούν ε, κατά την κατάρτιση αυτής της ετήσιας έκθεσης για τον παγκόσμιο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και αποτελεί και ένα πολύ σημαντικό βήμα ε, στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης συζητητέ για την ε, πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ε, έγιναν κάποιες δύσκολες συζητήσεις, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό για μένα. Προσπάθησα να λάβω υπόψη όλες τις πιθανές τροπολογίες κατά την διατύπωση των ε, τροπολογιών. Κάποιες τροπολογίες ήταν πολύ αναλυτικές και επικεντρώνονταν πάρα πολύ στις καθημερινές δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών και επομένω δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτή την έκθεση. Έκθεση η οποία αναφέρεται στις αρχές, στα θεσμικά όργανα και στις μείζονες μεταρρυθμίσεις ε, του ε, συστήματος των Ηνωμένων Εθνών. Σε ξεχωριστές τροπολογίες αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία ε, αρμόζουν στη φύση και στο πεδίο εφαρμογής της έκθεσης. Δεν μπορούσα βέβαια να συμπεριλάβω όλες τις τροπολογίες. Είχαμε 322 τροπολογίες. Ο κατάλογος ε, ψηφοφοριών ε, είναι έτοιμος και ελπίζω ότι αύριο θα διεξαχθεί ομαλά η ψηφοφορία. Ε, είχα πολύ καλή βοήθεια από τη γραμματεία της Επιτροπής και θεωρώ ότι τα πάντα έχουν προχωρήσει καλώς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια και ερωτήσεις. Uh, Ευχαριστώ κύριε Βοράινεν. Θα σας κάνω και εγώ την παρουσίαση εκ μέρους του κυρίου από το ΕΛΚ, αλλά θα δώσω πρώτα το λόγο στον Γιώ. Äh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι ο αλλά θα μιλήσω σαν μέλος ε, της ε, ομάδας εργασίας εδώ στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποτάσεων. Νομίζω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο αριθμός των τροπολογιών δείχνει ότι ουσιαστικά όλοι κοιτάμε προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να λάβουν χώρα στα Ηνωμένα Έθνη και βεβαίως ε, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών έδωσε μια όθηση σε αυτές τις εργασίες. Κοιτάμε προς το μέλλον, κοιτάμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την παγκόσμια διακυβέρνηση. Τον 21ο αιώνα η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα εδώ να μην σκεφτούμε ότι δίπλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας πρέπει να υπάρχει ένα Συμβούλιο Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, αυτό το ECOSOC. Και ο εισηγητής πολύ σωστά είπε ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταρρυθμιστεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι είπε ο εισηγητής. Νομίζω το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για το ΕΚΟΣΟΚ. Το θέμα της βιωσιμότητας όμως σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχυθεί η πτυχή βιωσιμότητα και η δημοκρατική πτυχή της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Βεβαίως τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα σύνολο κρατών με τις κυβερνήσεις τους. Εμείς σήμερα οφείλουμε να στοχεύσουμε στην καθημερινότητα των πολιτών και βεβαίως περισσότερη δημοκρατική, αν θέλετε, συνιστόσα μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Εμείς εδώ είμαστε ένα κοινοβούλιο. Εκπροσωπούνται πολλά διαφορετικά κοινοβούλια. Και βεβαίως τα παγκόσμια θέματα, τα θέματα που μας αφορούν όλους, είναι θέματα που θα πρέπει σίγουρα να συμπεριλαμβάνονται στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το θέμα του περιβάλλοντος και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά είναι θέματα παγκόσμια που αφορούν την ανθρωπότητα και που αποτελούν την καρδιά της πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. ο κύριος Μποστινάρο, ο οποίος θα μιλήσει εξ ονόματος του σκιώδους ε, των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσίαση αυτού του θέματος, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ξανά δει ότι οι πολύ σημαντικοί ηγέτες είχαν ε, σκεφτεί τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών σε μεγάλες διαφορές, σε μεγάλες συγκρούσεις και διαμάχες. Και νομίζω ότι σήμερα εν ώψη των πολλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε, ο ρόλος αυτός ε, είναι καθοριστικός, ε, καθώς και ο δικός μας. Θα μιλήσω λοιπόν εδώ εξ ονόματος του των σοσιαλιστών η οποία έχει καθυστέρηση στην ε, πτήση της. Καταρχήν χαιρετίζει το εξαιρετικό πνεύμα στο οποίο έλαβαν χώρα αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά το νέο Συμβούλιο για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε εδώ σε μια συμβαστική λύση. Υπάρχει η δομή και το σύστημα των ε, Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει εμείς να ενισχύσουμε εδώ το ΕΚΟΣΟΚ, χωρίς όμως να αποκλείσουμε την πιθανή του εξέλιξη μετεξέλιξη στο μέλλον. Πολλές, πολύ σημαντικές ε, τροπολογίες έχουν υποβληθεί από διάφορες ε, πολιτικές ομάδες όσον αφορά τη διαφάνεια στην εκλογή του Γενικού Γραμματέα και να υπάρχει βεβαίως ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε αυτήν την θέση. Συμβαστική τροπολογία 2 και εδώ ομιλούμε για τις ίσες ευκαιρίες και την ε, εξάλληψη των διακρίσεων από το 1945 δεν υπήρξε ποτέ γυναίκα Γενικός Γραμματέας. Και βεβαίως εδώ κοιτάξτε και τι προβλέπει το ψήφισμα 1321. Υπάρχει επίσης και η τροπολογία που δείχνει την δέσμευση την δική μας αναγνωρίζουμε το ρόλο που μπορεί να παίξει μια γυναίκα στην επίλυση διαφορών και στην βιώσιμη επίτευξη της ειρήνης. Πρόκειται και εδώ για μία από τις συμβαστικές τροπολογίες που θέλουμε σε κάθε περίπτωση να στηρίξουμε. Τροπολογία 203, δικαιοστάσιο όσον αφορά την θανατική ποινή και τις εκτελέσεις. 203 επαναλαμβάνω, η τροπολογία 203, η τροπολογία 205, οι λεγόμενοι κλιματικοί πρόσφυγες, ο ορισμός, καθώς και ο νομικός ορισμός, καθώς και δεσμευτικές, νομικά δεσμευτικές συμφωνίες. Θα θέλαμε πολύ να μπει αυτή η πρόταση μέσα στην συμβιβαστική τροπολογία, καθότι είχε οθετηθεί από την ετήσια έκθεση νωρίτερα το 2015. Ελπίζω ότι για την τροπολογία αυτή 205 θα υπάρξει πλειοψηφία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι στις ομιλίες πολλών ηγετών στην ε, ετήσια συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρθηκε ο όρος κλιματικοί πρόσφυγες. Φυσικά καθότι έχουμε μπροστά μας μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση, ίσως τη σοβαρότερη την οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Ανταπτυγκού έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Κιόδους, γιατί πραγματικά υπήρχαν πολλές τροπολογίες, πολύ διαφορετικές τροπολογίες και η προσπάθεια αυτή να φτάσουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες, σε κοινά κείμενα, είναι πολύ σημαντική για την συμπλήρωση και τον εμπλουτισμό αυτού του κειμένου. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ συγκεκριμένος ότι πρέπει να εξελιχθεί και ότι βεβαίως έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία μετάβασης, μεταρρύθμισης. Εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε και με την έκθεση αυτή δείχνουμε ποια θα μπορούσε να είναι η κατεύθυνση, ποιες θα πρέπει να είναι οι μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο στο γενικότερο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και της Γενικής Συνέλευσης, του Κοινικού Γραμματέα και βεβαίως ε, πώς μπορούμε και εμείς ε, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρουμε σε μια πιο αποτελεσματική εργασία. Προσπαθήσαμε με τις τροπολογίες μας να δείξουμε ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να ενσωματωθούν κάποια από τα δικά μας σημεία στις ήδη ενεξελίξει μεταρρυθμίσεις, αυτές δηλαδή που έχουν ξεκινήσει. Και θεωρώ ότι και μετά την Γενική Συνέλευση, την ετήσια Γενική Συνέλευση και αυτά που ακούστηκαν, βλέπουμε ότι θα μπορούσε σίγουρα η δημοκρατία, η βιωσιμότητα να αποτελέσουν πιο δυνατές πτυχές αυτού του οργανισμού. Δεύτερον, όπως ακριβώς ε, και ο Γιώ Λάινεν, θα ήθελα και εγώ να πω ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές τροπολογίες που ενισχύουν αυτήν την δημοκρατική πτυχή ε, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Ξέρουμε ότι σήμερα υπάρχουν εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι εκφράζουν δυσπιστία όσον αφορά την κυβέρνηση των χωρών τους. Όμως τα Ηνωμένα Έθνη εκπροσωπούνται από τις κυβερνήσεις τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν όλους αυτούς τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να ενισχυθούν, να ενισχυθεί ο ρόλος τους έτσι ώστε αυτή η δημοκρατική πτυχή του ΟΗΕ να ενισχυθεί. Μία πιο ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση επίσης. Ξέρω ότι αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ περίπλοκο, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Και αναφέρομαι εδώ στην τροπολογία 36. Η κοινωνία των πολιτών σίγουρα θα πρέπει να παίξει έναν πιο ισχυρό ρόλο στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Και πιστεύω ότι η τροπολογία αυτή θα υποστηριχθεί από εσά. Τώρα, όσον αφορά την εκλογή του Γενικού Γραμματέα, ίσως θα έπρεπε να ήμασταν λίγο πιο τολμηροί εδώ. Περιμέναμε κάτι παραπάνω από τον εισηγητή. Πραγματικά εδώ χρειάζεται αλλαγή έτσι ώστε να υπάρξουν νέες προτάσεις. Η συμβιβαστική 2 είναι σημαντική, πάει στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ίσως θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο τολμηροί. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να έχουμε το φάρος. Ξέρω ότι εδώ δεν συμφωνούν όλες οι πολιτικές ομάδες ε, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω έτσι ώστε να υπάρχουν γυναίκες αυτές τις θέσεις, περισσότερες γυναίκες. Νομίζω όμως ότι όλες αυτές τις συμβαστικές προτάσεις ε, ε, ενισχύουν προς τη σωστή κατεύθυνση το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την κούρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συνάδελφους στην Πάπερα Λακουίτου. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία. Και επειδή πάρα πολλέ ε, από τι ε, τροπολογίε μα ελήφθησαν υπόψη στου συμβιβασμού, θα ήθελα να αφαιρεθώ σε κάποιε τροπολογίε που δεν καλύπτονται από του συμβιβασμού, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικέ για τι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένων Εθνών η τροπολογία 167 για μια ευρωπαϊκή έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ε, αυτό θα ενίσχυε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή και θα αντικατοπτριζόταν ο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκοσμιο παίκτη. Ήταν δύσκολο να το πετύχουμε, αλλά νομίζω πρέπει να ασκήσουμε πίεση. Επίσης, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είμαστε η μόνη περιοχή στον κόσμο που έχει το δικαστήριό τη και έχει δικαιοδοσία επί των εθνικών δικαστηρίων και μπορούν σε αυτό να προσφύγουν και οι πολίτες. Το δικαστήριο αυτό έχει συνεισφέρει τα μάλα για ε, τον σεβασμό και την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και για άλλες περιοχές φαινομένα έθνη και κατόπιν ερευνευτικές αποστολές. Ε, μόλις το Σεπτέμβριο οργανώθηκε μια συνόδος κορφής ε, για το θέμα αυτό και πολλές χώρες όπως η Κίνα έχουν δεσμεύσει προς τα στρατεύματα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν περισσότερα στο θέμα αυτό. Επίσης ε, για τη χρήση των ντρόν, των μη αεροσκαφών, τροπολογία 299, τονίσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να έχουμε μία αυστηρή ερμηνεία ενός διεθνούς ε, νομικού πλαισίου που θα ορίσει ότι η χρήση των ενοπλών ντρόν θα πρέπει να σέβεται τη διεθνή νομοθεσία. Και τέλος, τροπολογία 300 για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αν πιστεύουμε στο ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τα Ηνωμένα Έθνη και το διεθνές δίκαιο, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μην παρεμβαίνουν στρατιωτικά χωρίς την εντολή των Ηνωμένων Εθνών. επομένω, θα πρέπει να υπενθυμηθεί στα κράτη-μέλη η δέσμευσή του για το διεθνές δίκαιο, ότι δεν θα πρέπει λοιπόν να παρεμβαίνουν στρατιωτικά, να παίρνουν στρατιωτικά χωρίς εντολή από τα Ηνωμένα Έθνη και να μην γίνεται παραβίαση της χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές λοιπόν είναι πολύ σημαντικές για μας και ελπίζω κατά την αυρινή ψηφοφορία να υπάρχει υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λοχμπίλερ. Ο κύριος Κάρφερ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα σας επιλέξει να ακούσετε ότι δεν μπορώ να συμφωνήσω. Γιατί ε, ουσιαστικά δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι να δοθεί μεγαλύτερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί των ε, κρατών μελών. Είδαμε, ε, ξέρετε εδώ ότι έχουμε δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη τη Γαλλία και τον Μένο Βασίλειο που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Φυσικά δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που προτείνεται και επομένως αναμένω την έντονη συζήτηση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να έχουν ζητήσει το λόγο. Έτσι λοιπόν θα κάνω και εγώ κάποια σχόλια του κυρίου Ντανζέν, του εισηγητή του ΕΛΚ που δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα, ο οποίος εκτίμησε τη στενή συνεργασία που είχε με τον εισηγητή, τον κύριο Βαράινεν και είναι ικανοποιημένο από τις κοινέ προσπαθίες σας που κατέληξαν σε ένα κείμενο το οποίο τώρα είναι ευρέως αποδεκτό από όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στο εγχείρημα αυτό. Ιδίω ε, είμαι ικανοποιημένο που επικεντρώνεται τώρα η έκθεση περισσότερο στην ε, στρατηγική για τις εξωτερικές υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ότι ουσιαστικά τώρα δίνουμε τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επικεντρωνόμαστε τόσο στην διακυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, ε, κατανοεί τις ε, προσπάθειες ε, του εισηγητή προς την κατεύθυνση του να δημιουργηθεί αυτό το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης και βλέπω τη διατύπωση που έχετε βρει ως συμβιβασμό φαίνεται να είναι κατάλληλη για όλους. Επίσης, τώρα η δομή της έκθεσης είναι πολύ ισορροπημένη μεταξύ της αιτιολογικής σκέψης και του κυρίως μέρους του κειμένου και η τεχνική διατύπωση είναι τώρα πιο ακριβής σε ό,τι αφορά ε, το ρόλο του, είπα, το, της, εξωτερικέ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξωτερικές υποθέσεις. Επίσης, ο κ. Στανσόν μπορεί να συμφωνήσει με τα περισσότερα αποτελέσματα στους 24 συνδεσμούς. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με ένα, αλλά νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για το αν θα αναφέρεται στο πώς θα πρέπει να γίνεται ακριβώς η διαδικασία του Γενικού Γραμματέα. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε ισορροπία μεταξύ των δύο φέλιων, ποτέ δεν είχαμε μία γυναίκα γενικό γραμματέα μέχρι τώρα αλλά αυτό είναι κάτι που πιστεύουμε ότι ίσως ε, θα έπρεπε να αποφασιστεί από τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι τα κυρία σχόλια του κύριου Ντάνζο. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, ίσως να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή για να συνοψίσει τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Θα είμαι σύντομος. Σημείωσα όλες τις επιθυμίες που εξακολουθείτε να έχετε και την υποστήριξη που εκφράσετε στις ατομικές σας τροπολογίες. Από ό,τι κατάλαβε, περισσότερες ομάδες υποστηρίζουν τώρα τις συμβαστικές τροπολογίες και από την πρώτη του ΕΛΚ υπάρχει κάποιος δισταγμός, κάποιες επιφυλάξεις για τη συμβαστική 2. Μπορεί να καταψηφίσει το ΕΛΚ, θα δούμε αύριο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Όμως, ε, αν δω εδώ τον κατάλογο ψηφορίας και δικές μου συστάσεις, θα γίνει κάποια αναθεώρηση και βάση της συζήτηση που είχαμε. Βλέπω ότι είμαστε όλο ένα και πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Αποτελεί λοιπόν αυτή μια καλή βάση για να οικοδομήσουμε τις θέσεις μας στο μέλλον. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλέ ιδέε που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια τέτοια έκθεση. Αν υπάρχει ένα πλήν, ω δική μου ένδειξη, για κάποιε τροπολογίε, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακή ιδέα ή ότι δεν συμφωνώ. Όμως, σημαίνει ότι η δομή της έκθεση και η φύση της έκθεσης περιορίζεται ότι μπορώ να δεκτώ εγώ. Βέβαια, στην, ψηφοφορία θα αποφασίσει πλειοψηφία και θα καθοριστεί έτσι το τελικό αποτέλεσμα. Α επικεντρωθούμε λοιπόν στην αυριανή ψηφοφορία και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια έκθεση λογική και θα έχει και μια δομική ενότητα. Και θα ακολουθεί τις αρχές που προσπάθησα εγώ να ακολουθήσω στο, δική μου, στο δικό μου σχέδιο έκθεση όταν διαπραγματευόμασταν τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βερένεν, ευχαριστούμε και τους Κιώδης. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το θέμα στην σε διάταξη και υπενθυμίζω ότι αύριο θα ψηφίσουμε στις 10 παρατέταρτο. Όλοι αναμένετε να συμμετέχετε αύριο στην ψηφοφορία μετά τη συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Ο κύριος Κρίστιαν Λέφλερ, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα τη Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα έρθει σε λίγο. Μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Και θα ξεκινήσουμε στις 4 και πάλι. Okay, dear colleagues, uh, Λοιπόν, συνάδελφοι, πήγε τέσσερις. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το σημείο πέντε της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Κρίστιαν Λέφρεν, τον οποίον καλωσορίζω θερμά. Είναι ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για οικονομικά και παγκόσμια ζητήματα. Ήταν πριν ε, διευθύνων σύμβουλος. Τώρα είναι πρώτη φορά εδώ με τη νέα του ιδιότητα. Καταρχάς να σας πω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κούβας απολαμβάνουν μια όθηση χωρί προηγούμενο. Υπάρχουν διαπραγματεύσει για την ολοκλήρωση πολιτικού διαλόγου και συμφωνία συνεργασία. Να έχουμε λοιπόν μια εταιρική σχέση. Η Κούβα είναι η μόνη χώρα τη Λατινική Αμερική που δεν έχει συνάψει συμφωνία ε, συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση για προφανείς λόγους βεβαίως όπως όλοι γνωρίζουμε. Εκ παραλλήλου, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, της Αμερικής και η Κούβα αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές του σχέσεις την 1η Ιουλίου του 2015 και όλοι ε, υπήρξαμε μάρτυρες αυτής της ιστορικής επαναπροσέγγισης μεταξύ των ε, δύο χωρών η οποία είχε ξεκινήσει από τα τέλη του προηγούμενου έτους. Βέβαια, για να εξομαλυνθούν πλήρως ε, οι σχέσεις, ε, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο. κυρίως λόγω του οικονομικού εμπάργου των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας. Ε, τον Ιούνιο του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ξεκινήσει ένα πλήρη πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση της Κούβας. Έκτοτε έχουν γίνει έξι ε, συναντήσεις υψηλού επίπεδου σε πολιτικό επίπεδο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί σχέσεις με την Κούβα εδώ και 27 χρόνια και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο ανέκαθεν ήταν ε, βήμα διαλόγου. Οι Ευρωβουλευτές ήταν σε επαφή με κουβανούς εταίρους από το 1995. Έχουμε λοιπόν περίπου 30 χρόνια διαλόγου και Ε, είχαμε σχέσεις με το Παρλατίνο που έχει και κουβανούς ε, βουλευτές. Το Δεκέμβριο του 1996 ξεκίνησε η σχέση συνεργασίας και θέλουμε να έχουμε μια μετάβαση προς μια πολυφωνική δημοκρατία, καθώς επίσης να υπάρχει και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελωδιών ελευθεριών. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα μας δίνει τη ευκαιρία να δούμε πώς ε, αξιολογεί την πρόοδο που επιτελεί η Κούβα τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τι ε, μέλη γενέστε για τον πολιτικό διάλογο και τη συμφωνία συνεργασίας και επειδή ο κύριος Λέφλερ επισκέφθηκε την Κούβα τον περασμένο μήνα, θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια για τις ε, πιο πρόσφατες εντυπώσεις του, για το πώς ε, αντιμετωπίζει η χώρα αυτό το νέο μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο έχει βρεθεί. Επίσης θα θέλαμε να ακούσουμε και κάποια σχόλια για την πρόσφατη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Κούφα καθώς επίσης και τις βασικές οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και γενικότερα την κοινωνική και οικονομική κατάσταση της χώρας, δεδομένου ότι ήταν απομονωμένη για τόσα χρόνια. Αυτά λοιπόν εισαγωγικά από πλευρά μου και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Λέφλερ να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μου δίνεται πολύ δύσκολο καθήκον Πράγματι, για πρώτη φορά έρχομαι στον Μερκοβουλίο υπό ε, αυτές τις ε, αρμοδιότητες, αλλά είχα ξανάρθει να μιλήσω για την Κούβα ως διαπραγματευτής της ε, συμφωνίας ε, με την Κούβα και επομένως έχω ξανάρθει στο παρελθόν για να μιλήσω για το θέμα αυτό. Και πράγματι, συζητήσαμε το θέμα της Κούβας και στην ε, Ολομέλεια τον Ιούλιο, όπου ο Επίτροπος Χαν και είπατε πρόσωπος ε, συζήτησαν ε, θέματα που είχαν να κάνουν με τη σχέση με τη Λατινική Αμερική και με την Κούβα. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί για την κατάσταση στη χώρα και για τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας ε, είναι η αλλαγή και η συνέχεια. Εγώ τώρα δεν θα πω ε, συνέχεια και αλλαγή, θα τα πω αντίστροφα. Υπάρχει αλλαγή στις σχέσεις μας, υπάρχει αλλαγή στην Κούβα και φυσικά υπάρχει και αλλαγή στο συνολικό πλαίσιο, στο πώς εξελίσσεται η Κούβα, ιδίω στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι ισχυροί παράγοντες συνέχειας υπάρχει και μια μεγάλη βούληση από την κουβανική ηγεσία να διατηρήσει ένα υψηλό βαθμό συνέχειας στις δομές και στις πολιτικές τους. Και βέβαια κάτι τέτοιο δεν ε, ακολουθεί πάντοτε τους ε, στόχους ε, που έχουν κάποιοι εταίροι τους παγκοσμίως. Η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή τον τελευταίο χρόνο είναι σαφώς η προσέγγιση μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κούβα βγήκε από την απομόνωση στην Αμερικανική Ήπειρο και αυτή η απομόνωση ήταν πάντοτε σχετική, όμως ε, το περασμένο έτος, είστε λιγότερο από ένα έτος, δηλαδή από πέρσι το Δεκέμβριο, η Κούβα έχει αναδυθεί ως ένας ισχυρός και ενεργός περιφερειακός παίκτη και μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε ε, συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα όπως είδαμε και στη διάσκεψη της Αμερικανικής Επίρου. Και έχουν ε, αναλάβει έναν ισχυρό ρόλο στην διεθνή σκηνή με την επίσκεψη του Φραγκίσκου το Σεπτέμβριο. Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη ΠΑΠΑ στην Κούβα τα τελευταία 20 χρόνια. Και νομίζω ότι ήταν επιτυχής η επίσκεψη αυτή και για την Κούβα και για τον ΠΑΠΑ. Η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, η εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, ε, αν και ίσως ε, δεν έχει γίνει ακόμα εξομάλυνση σε οικονομικό επίπεδο, και η ενδυνάμει ανάπτυξη του αμερικανικού τουρισμού στην Κούβα και στις σχέσεις μεταξύ των δύο έχει σημειώσει αύξηση πάνω από 20% τους τελευταίους δύο μήνες. Όλα αυτά αλλάζουν το τοπίο στη χώρα. Αυτό είναι και εμφανές, αλλά αλλάζουν και οι προσδοκίες σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Αυτή είναι μια πρόκληση για μας, αλλά είναι και υποστήριξη στις δικές μας προσπάθειες να επιδιώξουμε και να αναπτύξουμε και να εμβαθύνουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας. Όπως γνωρίζετε, αυτό το πράττουμε αρκετά χρόνια. Όπως αναφέρεται, το 2008 όταν μετά από κάποια έτη διακοπής του πολιτικού διαλόγου και της οικονομικής συνεργασίας, αυτά ξαναξεκίνησαν, υπήρξε νέα ανάληψη δέσμευσης και μετά από κάποια χρόνια διαλόγου, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβαν την πρωτοβουλία να προτείνουν στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο για τις σχέσεις μας και να διαπραγματευτούμε ένα πολιτικό διάλογο και συμφωνία συνεργασίας μετακινούμενοι από ένα χαλαρό άτυπο πλαίσιο σε μια ισχυρή νομική μορφή που είναι ο πολιτικός διάλογος και συμφωνία συνεργασίας. Θα γνωρίζετε ότι οι κουβανικές αρχές για πολλά χρόνια, για 20 χρόνια, έβλεπαν ε, ως αγκάθι την ευρωπαϊκή κοινή θέση. ως ε, μονομερή ε, δήλωση πρόθεσης από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ουσιαστικά πρόκειται για μια τέτοια μονομερή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όσους έχετε παρακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό την ευρωπαϊκή πολιτική θα θυμάστε ότι η ιδέα των κοινών θέσεων, το μέσο αυτό αποτελούσε ένα πείραμα της συνθήκης του Άμστερνταμ και κάποιες ε, είχαν υιοθετηθεί νομίζω μόνο μία κοινή στρατηγική υπήρχε τότε. Οι περισσότερες ε, είτε εξαφανίστηκαν είτε λησμονήθηκαν. Και μία μόνο έμεινε και ήταν η κοινή θέση απέναντι στην Κούβα. Και ουσιαστικά δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ήταν αυτό το μόνο που είχαμε. Και απόφαση που ελήφθη πριν λίγα χρόνια να προτείνουμε να προχωρήσουμε σε μια συμφωνία πλαίσιο ανταυτού βασίστηκε στην πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος να δώσουμε όθηση στην αλλαγή και στην ανάπτυξη στην Κούβα είναι να συνεργαστούμε μαζί τους και να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους σταθερούς τρόπους να το κάνουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα όπου έχουμε διαφορετικές οπτικές, όπου διαφωνούμε. Όμως αυτό συμβαίνει με πάρα πολλές χώρες στον κόσμο και δεν υπάρχει λόγος να μην συνεργαστούμε. It's on that basis. Βάσει αυτού, ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις ε, για το νέο πλαίσιο συνομιλιών, οι οποίες ε, βρίσκονται εν εξελίξη ξεκίνησαν πριν από 1,5 χρόνο και ο πέμπτος ε, γύρος ε, συζητήσεων έλαβε χώρα στην Αβάνα το Σεπτέμβριο, ήμουν παρόν και ο επόμενος γύρος θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό ίσως σας φανεί σαν ε, μια διαδικασία που αργεί. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Προσπάθησα να συγκρίνω το πλαίσιο των συζητήσεων για τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Και πραγματικά, όπως ξέρετε, με τον Καναδά έχουμε πολλά κοινά σημεία. Δεν ήταν ένας δύσκολος εταίρος. 13 γύρι συνομιλιών έλαβαν χώρα. Και εδώ είμαστε στο δεύτερο χρόνο και στον πέμπτο γύρο με την Κούβα. Άρα τα πράγματα βαίνουν καλώς, έχει επιτευχθεί πολύ σημαντική πρόοδος και βασιζόμαστε για αυτή τη συμφωνία σε τρεις πυλώνες. Πολιτικός διάλογος που συμπεριλαμβάνει σημαντικά πολιτικά θέματα, πολυμερή συνεργασία, περιφερειακή συνεργασία, διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα. θεμελιώδη οικονομικά, κοινωνικά δικαιώματα και βεβαίως κάποιες διεθνείς προκλήσεις, μετανάστευση, ναρκωτικά, βιώσιμη ανάπτυξη, διακρίσεις κτλ. κτλ. Και άλλα θέματα πιο παραδοσιακά που εμπίπτουν στην εξωτερική πολιτική, τα όπλα μαζικής εξάλληψης κτλ. κτλ. Τα άλλα δύο κεφάλαια, οι άλλοι δύο πυλώνες είναι ο ένας έχει τίτλο «Συνεργασία και διάλογος που αφορά την πολιτική», συμπεριλαμβάνει την γεωργία, το περιβάλλον και άλλα θέματα. Θέλουμε να δημιουργηθεί διάλογος μεταξύ εμπειρογνωμόνων, μεταξύ ειδικών, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένους τομείς, στους οποίους μπορεί να υπάρξει συνεργασία, αφού προηγουμένως έχουμε εξετάσει τους τομείς αυτούς. Ο τρίτος πυλώνας είναι οι οικονομικές σχέσεις. Δεν πρόκειται για προτιμησιακή συμφωνία. Δεν πρόκειται για συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ούτε προτιμησιακών εμπορικών συναλλαγών. Αυτό είχε ζητήσει η Κούβα. Εδώ πρόκειται ουσιαστικά για κάποιες, αν θέλετε, εγγυήσεις ότι ερμηνεύουμε με τον ίδιο τρόπο τους διεθνείς κανόνες, τα διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να συνεργαστούμε για θέματα προτύπων, για θέματα εμπορικά, έτσι ώστε να ενισχυθεί η τελωνιακή συνεργασία, θέματα που αφορούν ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο, τα διοικητικά θέματα, για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Τώρα, τα οικονομικά θέματα, θέματα συνεργασίες έχει προοδεύσει πολύ στον τομέα αυτό η συζήτηση. Και αν θέλετε τα δύο αυτά κεφάλαια σε μεγάλο βαθμό έχουμε σε μεγάλο βαθμό συμφωνήσει όσον αφορά τους όρους που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την σύναψη αυτής της συμφωνίας ε, πλαίσιο. και βεβαίως ε, όταν το κείμενο ετοιμαστεί θα υποβληθεί πρώτον στους πολιτικούς ηγέτες, κατόπιν ε, στο κοινοβούλιο εδώ και αντιστοίχως ε, στις αρχές της Κούβας. Όσον αφορά τον πολιτικό διάλογο, σε αυτό το πυλώνα, σε αυτό το κεφάλαιο επίσης έχει επιτευχθεί πρόοδος, παρόλα αυτά παραμένουν κάποια σημεία προς επεξεργασία, προς διευκρίνηση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι όταν προετοιμαστεί το τελικό πλαίσιο διαλόγου για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διακυβέρνησης, κατανοούμε με τον ίδιο τρόπο για ποιο διάλογο ομιλούμε. Ποια είναι τα όρια, μέχρι πού μπορούμε να δεσμευτούμε και πέρα από τις διαπραγματεύσεις αυτές καθεαυτές έχουμε ήδη ξεκινήσει μια άσκηση στον τομέα αυτό του πολιτικού διαλόγου πριν από το καλοκαίρι και ο Σταύρος Λαμπρινίδης πέρνος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ξεκίνησε έναν διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τον ε, ομολογό του, τον Υπουργό Εξωτερικών της Κούβας, ο Σταύρος και εγώ, είχαμε μια ολόκληρη μέρα διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και βεβαίως ε, δεν συμφωνήσαμε σε όλα τα θέματα τα οποία θίξαμε. Παρόλα αυτά νομίζω ότι έχει βρεθεί πολύ ε, σημαντικός χώρος συνεννόησης για τα περισσότερα σημεία τα οποία θίξαμε και στα οποία ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Ελπίζουμε ότι στον επόμενο γύρο που θα λάβει χώρα όπως σας είπα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου εδώ στις Βρυξέλλες και το 2000 στους επόμενους γύρους συζητήσεων που θα ακολουθήσουν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε πλήρη συμφωνία ή σχεδόν πλήρη συμφωνία και να ολοκληρώσουμε αυτόν τον πολιτικό διάλογο με την Κούβα. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι από τεχνικής απόψεως τουλάχιστον αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν βεβαίως η πολιτική βούληση συνεχίσει να υπάρχει. Από την πλευρά τη δική μας τουλάχιστον υπάρχει και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, να φτάσουμε στη θέσπιση αυτού του πλαισίου, έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η συνεργασία και οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Κούβα σαν μια σταθερή καθότι αυτή τη στιγμή η Κούβα αλλάζει και βεβαίως το βασικό καθοριστικό θα έλεγα στοιχείο αυτής της μεταρρύθμισης, αυτής της αλλαγής είναι οι νέες σχέσεις της Κούβας με τον μεγάλο γειτονά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Ομπάμα αναφέρθηκε όπως ξέρετε στο εμπάργο των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κούβα λέγοντας ότι είναι απαρχαιωμένο, ότι είναι αντιπαραγωγικό και ότι πρέπει φυσικά να πάψει να ισχύει. Εμείς συμφωνούμε, το πιστεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο εμποδίζει τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας, αλλά εμποδίζει και την οικονομική ανάπτυξη της Κούβας. Θέλουμε λοιπόν να συνεισφέρουμε σε αυτό, θέλουμε να βοηθήσουμε τον εξυγχρονισμό της Κούβας και φυσικά το εμπάργο εμποδίζει κάτι τέτοιο. Και φυσικά έχει πάρα πολύ αρνητικές ε, ε, ε, πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις συγγνώμη, στις σχέσεις μεταξύ Κούβας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε λοιπόν υπέρ της άρσης του εμπάργου. Η Κούβα βεβαίως έχει δραστηριοποιηθεί γενικότερα στην Νότια, στη Λατινική Αμερική και είναι ένας εταίρος στην Καραϊβική για άλλες μικρές χώρες. Είναι ένας σταθεο, σταθεροποιητικός παράγοντας για όλη την περιοχή της Δυτικής Αφρικής με την ιατρική της στήριξη. Πιστεύουμε ότι εκεί, σε αυτές τις αποστολές, μπορούμε να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε με την Κούβα έτσι ώστε να ενισχύσουμε τις επαφές μας, τις διμερείς επαφές μας με την Κούβα. Ανανεώσαμε λοιπόν και ενισχύσαμε το πρόγραμμα συνεργασίας μας με την Κούβα μέχρι το 2020 50 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός. Βεβαίως δεν είναι σημαντικός ε, προϋπολογισμός αν το συγκρίνει κανείς με άλλους προϋπολογισμούς συνεργασίας με άλλες χώρες, αλλά βεβαίως αν το συγκρίνει με τα ποσά που αφορούν την Κούβα σε σχέση με άλλα προγράμματα συνεργασίας στον κόσμο, είναι ένα σημαντικό ποσό θέλουμε να στηρίξουμε, να συνοδεύσουμε τις ε, πρωτοβουλίες συνεργασίας όσον αφορά την τεχνογνωσία, την εμπειρογνωμοσύνη, τον εξυγχρονισμό της μεταρρυθμίσεις στην Κούβα. Βεβαίως συνεχίζουν να υπάρχουν δυσκολίες στη χώρα και Υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες όσον αφορά θεμελιώδεις ελευθερίες, την ελευθερία του συνέρχεσθε, η ελευθερία έκφρασης. Πρόκειται για θέματα τα οποία συνεχίζουν να δυσκολεύουν ε, τις σχέσεις μας με την Κούβα. Και κάθε φορά που συναντάμε τους εταίρους μας, φύγουμε τα θέματα αυτά τα αναφέρουμε και τους έχουμε παροτρύνει τα τελευταία χρόνια να περάσουν από την υπογραφή των, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στην κύρωση και κυρίως στην εφαρμογή. Βεβαίως ε, δεν είναι εύκολο να περάσει κανείς από την υπογραφή στην κύρωση, αλλά σίγουρα η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι σημαντική και νομίζω ότι εδώ και 7 χρόνια εκρεμεί το κείμενο στο Κοινοβούλιο της ε, Κούβας. 7 χρόνια δεν έχει κυρωθεί θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει και το θέμα αυτό, πώς θα βελτιωθεί η κατάσταση και στον οικονομικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα, αλλά και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των πολιτών. Πιστεύουμε ότι ο πολιτικός διάλογος είναι ένας τομέας που θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ο διάλογος είναι πολύ σημαντικός για να προχωρήσει η κοινωνία της Κούβας σε εξυγχρονισμό, σε περισσότερη εμπιστοσύνη. Χωρίς εμπιστοσύνη, χωρίς διάλογο, ο εξυγχρονισμός δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλουμε να συνεχίσουμε την συνεργασία μας με τους εταίρους μας από την Κούβα σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά όχι μόνο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε περισσότερο εξυγχρονισμό και ευημερία στο νησί. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Λέφλερ για την ε, πληρέστατη παρουσίαση των σχέσεων με την Κούβα. Τρεις συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο προς το παρόν. Ο κύριος Γκάλερ καταρχάς. Μίχαηλ. Ε, ε Ευχαριστώ κύριε Λέφλερ για την πολύ τεκμηριωμένη σας παρουσίαση. Μας ενημερώσετε πόσο έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις με θετικό τρόπο εκτιμάται το αποτέλεσμα. Είναι πολύ θετικό το ότι έχει ξεκινήσει διάλογος, συνομιλίες με σκοπό να υπογραφεί μια συμφωνία. Μιλήσατε για αλλαγή και για συνέχεια. Change and continuity. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευτυχής που οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κούβα επαναξεκίνησαν διπλωματικές σχέσεις. Και βεβαίως το θέμα των κυρώσεων θα έπρεπε να είχαν σταματήσει αυτές οι κυρώσεις εδώ και 25 χρόνια. Σε καμία περίπτωση η Κούβα δεν ήταν κίνδυνος και απειλή για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Από τότε ήδη λοιπόν έπρεπε να υπάρξει άρση. Εν πάση περιπτώσει Ξέρουμε ότι το καθεστώς έχει αλλάξει και μιλήσατε για συνέχεια όσον αφορά τις δομές και την πολιτική. Τελικά αυτό που είναι καθοριστικό, αν κατάλαβα καλά, είναι το θέμα της εξουσίας. Αν δηλαδή υπάρχει μία μονοπωλιακή κατάσταση όσον αφορά την εξουσία, αν υπάρχουν δυνατότητες για μία δημοκρατική μεταρρύθμιση, αλλαγή. Είναι η μόνη χώρα στη Λατινική Αμερική που στις εκλογές εμφανίζεται ένα κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να μην ξεχνάμε ποια είναι η θέση μας ήδη από το 1996. Θεωρώ ότι αν διαβάσουμε αυτά που είχαμε πει τότε, ισχύουν όλα και σήμερα. Ζητάμε εκδημοκρατισμό, όπως σε όλη την ε, Αμερικανική Ήπειρο. Το είχαμε πει και πριν από 25 χρόνια, νομίζω το λέμε το ίδιο και σήμερα, ότι θα πρέπει να ζητήσουμε από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μιλάτε για διάλογο, για συνεργασία, για θέματα που αφορούν τον κρατικό μηχανισμό. Τι θα λέγατε, μπορούμε να ζητήσουμε από την κυβέρνηση της Κούβας να μας δώσει ένα χρονοδιάγραμμα πώς σκέφτεται να προχωρήσει στον εκδημοκρατισμό της χώρας. Συγγνώμη, και στην ε, Ανατολική Γερμανία ε, το ίδιο καθεστώς υπήρχε, αλλά βλέπετε όλη η Λατινική Αμερική έχει περάσει σε πιο δημοκρατικές διαδικασίες. Από ολοκληρωτικά καθεστώτα πέρασαν σε δημοκρατικά. Λίγο πολύ. Πραγματικά λοιπόν πριν από 25 χρόνια είχαμε ζητήσει αυτό το κομμουνιστικό καθεστώς να γίνει δημοκρατικό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιες είναι οι προοπτικές, πώς βλέπετε τα πράγματα. Δεν έχετε την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή το καθεστώς στην Κούβα κοιτάει την ιδιωτικοποίηση της οικονομίας, αλλά Ξέρουμε ότι υπάρχουν παραδείγματο χάρη ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν αυτήν την ιδιωτικοποίηση, αγοράζουν ξενοδοχεία, εποφελούνται από τις δυνατότητες της οικονομίας, της αγοράς. Και βλέπουμε ότι η καθεστοτική αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει να λειτουργούν σαν επενδυτές. Εγώ δεν θέλω να δω μια ιδιωτικοποίηση προς όφελος των ίδιων. Μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία που θα δώσει δύναμη στους πολίτες είναι αυτό που ζητάμε και σε καμία περίπτωση το παλιό καθεστώς να ξεκινήσει με προνόμια και να είναι στην πρώτη γραμμή έτσι ώστε να επωφεληθεί από την απελευθέρωση της ε, οικονομίας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας έτσι ώστε οι νέες μας σχέσεις να είναι υγιείς. Νομίζω ότι ήμουν ο τέταρτος. Όχι. Το 1998 άρχισα να παρακολουθώ στενά τις σχέσεις της Κούβας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, καταλαβαίνω γερμανικά, απλώς δεν ακούω καλά, δεν ακούω καλά. Θα μιλήσω πιο δυνατά. Από το 98 λοιπόν ασχολούμαι με το θέμα αυτό των σχέσεων ε, με την Κούβα. Έχω επισκεφτεί το νησί και θυμάμαι ότι πρόκειται για κάποιες εξαιρετικές συνθήκες και περιπτώσεις που οδήγησαν ε, την ε, Κούβα σε κάποιες αλλαγές. Η επίσκεψη του Πάπα σίγουρα θα είναι μία από αυτές. Η τελευταία επίσκεψη του Πάπα ήσασταν παρόν κατά την επίσκεψή του. Και θέλω να μου πείτε μία-δύο εβδομάδες ε, μετά επανήλθαν τα πάντα όπως ήταν. Όσον αφορά τώρα τη συμφωνία πλαίσιο την οποία επεξεργαζόμαστε, ναι, εδώ και 1,5 χρόνο επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη συμφωνία και συζήτησα με μια ειδική, μια εμπειρογνώμονα στη Μαδρίτη πριν από λίγο καιρό για αυτό το θέμα και αναρωτιέμαι, ήμασταν προετοιμασμένοι εμείς η Ευρώπη όταν ξεκίνησε η συνεργασία μεταξύ Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών. Εσείς στις Βρυξέλλες ξέρατε κάτι, είχατε ακούσει κάτι ότι προετοιμάζεται αυτή η προσέγγιση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας. Για μας ποιες είναι οι συνέπειες. Κινδυνεύουμε για άλλη μια φορά να βρεθούμε πίσω από τους Αμερικάνους. Και να είναι η δικιά μας συμφωνία πραγματικά καθυστερημένη. Το εμπάργο και η άρση του εμπάργου από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς ε, και οι εκλογές αλλά και ε, οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρετε πολύ καλά ότι σε καμία περίπτωση το θέμα της Κούβας δεν θα μείνει εκτός της προεκλογικής εκστρατείας. Και αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι οι πραγματικές συνέπειες στην Κούβα. Η Μαριάντα Σαρνέζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι εδώ μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι για την ιστορική στιγμή που διανύουν οι σχέσεις είπα και Φυσικά φυσικά ε, έπαιξαν οι Αμερικανοί έναν ισχυρό ρόλο και ο Πάπας έναν ισχυρό ρόλο εμείς μπορούμε να ρωτηθούμε βέβαια Ευρωπαίοι αν ήμασταν παρόντες από κοντά από μακριά αυτή είναι η πρώτη ερώτηση το δεύτερο Πιστεύω ότι τώρα το μόνο ζήτημα που είναι ενώπιόν μας είναι το εξής. Πώς εμείς θα συνοδεύσουμε στην Κούβα στη διπλή της μετάβαση. Υπάρχει μια οικονομική μετάβαση που θα πρέπει να γίνει και μια δημοκρατική μετάβαση. Και αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή τη διπλή μετάβαση γιατί είμαι βεβαισμένη για το ότι πρέπει να προχωρήσουμε και προς τους δύο στόχους ταυτόχρονα και να κάνουμε κάποια βήματα προς ε, αυτούς τους δύο στόχους ταυτόχρονα. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι σκέφτεστε για αυτή τη διπλή στρατηγική, είναι δυνατή και κατά δεύτερον αν οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν την ίδια προσέγγιση που έχουμε και εμείς, είναι διαφορετική η προσέγγιση τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Σακοράφα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ρέφλερ, μετά τα μετά από τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε και οι οποίες δείχνουν ότι στις σημερινές κρίσιμες συνθήκες όπου οι ψυχροπολεμικές φωνές εντείνονται, η προσπάθεια για παραπέρα ανάπτυξη σχέσεων με το σοσιαλιστικό κράτος των εργατών και αγροτών της Κούβας αποτελεί απάντηση σε όσους συνεχίζουν να προτείνουν αδιέξοδες πολιτικές όπως είναι η επεμβάση, οι και το εμπάρκο. Ε, Θεωρώ ότι η Συμφωνία Συνεργασίας και Πολιτικού Διαλόγου, στην οποία αναφερθήκατε εκτενέστατα προηγουμένω, δίνει ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης σχέσεων ισότιμων μεταξύ των δύο μερών. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι μια μικρή χώρα που για πάνω από 50 χρόνια βιώνει την ε, πίεση ενός δολοφονικού εμπάρκου προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση ισότιμα. Γνωρίζοντας λοιπόν πολύ καλά την πολιτική και την οικονομική συγκυρία, ξέρω ότι αυτή η προσπάθεια θα χρειαστεί ιδιαίτερο κόπο φυσικά, αλλά και ανοιχτή αντίληψη από όλες τις πλευρές. Από την πλευρά μας νομίζω ότι οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι αυτή η κοινή προσπάθεια θα διέπεται από τις αρχές της χωρίς όρους και χωρίς διακρίσεις αμοιβαιότητας και συνεργασία. Και στο πλαίσιο αυτό επίσης πιστεύω ότι η επίσημη κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από το 1996, αποτελεί εμπόδιο για την ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, καθώς παραβιάζει την αρχή της μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών και στην πραγματικότητα είναι περιττή με δεδομένο ότι τα κράτη-μέλη έχουν ήδη συνάψει διμερείς σχέσεις με την Κούβα. Θέλω λοιπόν να ελπίζω ότι ο κοινό βηματισμό μα θα έχει γρήγορα μετρήσιμα και επωφελή αποτελέσματα για του λαού μα και από αυτή την άποψη θεωρώ ιδιαίτερα θετικό το γεγονό ότι οι μέχρι τώρα συζητήσει έχουν γίνει και έχουν διεξαχθεί σε επικοδομητικό περιβάλλον, δείχνοντα με τον τρόπο αυτό τη δέσμευση των δύο πλευρών να συνεχίσουν την ευάθυνση των σχέσεών του και να προχωρήσουν γρήγορα προ τη σύναψη τη συμφωνία στην οποία αναφερθήκατε. Όπω επίση προσωπικά θέλω να τονίσω ότι στηρίζω με όλε μου τι δυνάμει την παραπέρα ανάπτυξη των σχέσεων με την Κούβα, με απόλυτο σεβασμό σε ένα λόγο που ακόμα και κάτω από τι πιο αντίξωε συνθήκε κατάφερε να μην εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την αξιοπρέπειά του και το δικαίωμά του να αποφασίζει αυτό για τη ζωή του και τη χώρα του, ελπίζοντα φυσικά ότι στο επόμενο, στην επόμενη διαδικασία τη συζήτηση στα Ηνωμένα Έθνη όσον αφορά το θέμα του, του αποκλεισμού τη Κούβα, ε, ότι το αποτέλεσμα θα καταλήξει να είναι θετικό από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very Ευχαριστώ, κυρία Σακοράφα. Ο κύριος Μιλάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τον κύριο Λέφλερ και Καταρχήν να σας ε, πω συγχαρητήρια για το διορισμό σας ε, και την προαγωγή σας εντός της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Επίσης, ε, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μας κάνετε. Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι σε αυτή τη διαδικασία που ήδη κρατά ένα μισή χρόνο και έχουμε ήδη και τον πέμπτο γύρο διαπραγματεύσεων. Προσέξατε κάποια αλλαγή την ε, θέση της Κούβας ε, κυρίως ε, λόγω του νέου σκηνικού της εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει κάποιος αντίκτυπος. Εγώ υποθέτω πως ναι, απριόρι, αλλά εσείς που ε, έχετε από κοντά ε, δει και τα θέματα. Ποιες είναι οι προοπτικές ε, του να δημιουργηθεί μια πραγματική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας. Εγώ νομίζω ότι καθώς έχουμε την εξομάλυνση των σχέσεων της Κούβας με τις Πολιτείες αυτό θα έπρεπε να έχει και ένα αντίκτυπο στις σχέσεις που θα έχει η Κούβα με εμάς και βλέπετε ότι θα υπάρχει Κάποιο αντίκτυπος εκεί ή επειδή έχουν πετύχει αυτή την εξομάλυνση πιστεύετε ότι δεν θα έχουν τόσο πολύ ανάγκη για να συνάψουν και σχέσεις μαζί μας. Έχετε προσέξει λοιπόν κάτι, αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Δεύτερον, μου δίνεται η εντύπωση ότι από εμπορική πτυχή. Όπως είπατε δεν είναι προτιμησιακή συμφωνία, δεν έχει ιδιαίτερο περιεχόμενο ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά των προϊόντων. Από ό,τι κατάλαβα έχουμε βελτίωση των τελειωνιακών συστημάτων, ε, υπάρχει κάτι σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτόν τον οικονομικό πυλώνα της συμφωνίας. Τρίτον, εγώ βλέπω τη δική μας συμφωνία βασικά ως ε, ουσιαστικά μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει θέση έναντι μιας ε, μετάβασης, ανεπόφευκτης μετάβασης ε, στην Κούβα. Φυσικά θα υπάρξει αλλαγή, θα δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η μετάβαση. Η συμφωνία αυτή θέλει να ενισχύσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι πιο παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτούς ε, τους καιρούς ε, της αλλαγής του καθεστώτος ή της μη αλλαγής. Γιατί εσείς μιλήσατε για αλλαγή και συνέχεια. Εγώ πιστεύω ότι η ουσιαστική ε, φύση του καθεστώτος έχει κάπως τροποποιηθεί. Έτσι λοιπόν από αυτή την ε, οπτική θα ήθελα να θεστήσω την προσοχή σας ε, στο η σημασία έδινε το Κοινοβούλιο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ε, χαίρομαι που τέθηκε σε εφαρμογή αυτός ο διάλογος με τον επανταρμόστη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως θα ήθελα να ε, επισημάνω και σε πόσους ε, πολιτικούς αντιρρησίες της Κούβας έχει δοθεί το βραβείο Ζαχάροφ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Έτσι λοιπόν το σημαντικό είναι να έχει ένα περιεχόμενο ο διάλογος αυτός και αν εσείς μπορέσετε να έχετε και κάποια επιρροή στην ε, επικύρωση της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Φρονών για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την πλευρά της Κούβας, πόσο το καλύτερο. Εγώ νομίζω ότι ε, όμως με το πέρασμα του χρόνου και για βιολογικούς λόγους θα υπάρχει αλλαγή και στο πολιτικό κομμάτι του καθεστώτος. Τώρα, στο εμπάργκο στο οποίο αναφερθήκατε. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εσείς εκτιμάτε όλο αυτό το ζήτημα για το μέλλον. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο. Το θέμα του εμπάργου ε, δεν είναι στην αρμοδιότητα του Λευκού αλλά του Κογκρέσου. Και αν δεν αλλάξουν οι πλειοψηφίε στο Κογκρέσο, βλέπω δύσκολο να αλλάξει και το θέμα του εμπάργου. Θα θέλω ε, να μας πείτε πώς το βλέπετε εσείς, το ζήτημα αυτό και ποια είναι η εκτίμησή σας, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το ζήτημα από την πλευρά της Αμερικανικής Διοίκησης ή από την πλευρά του Κογκρέσου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μποστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεφλέρ για τη συνεισφορά σας ήταν πλήρης η παρουσίασή σας και ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα πόσο περίπλοκες είναι οι σχέσεις μας με την Κούβα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πρέπει να εξετάζουμε την, την Κούβα τουλάχιστον με τρεις διαφορετικές διαστάσεις. Καταρχάς, σε σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, συγγνώμη, Πολιτειών. είναι αλήθεια ότι παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση τα τελευταία χρόνια ε, με τη σχέση μας με την Κούβα. Μας εξέπλεξε ε, η όθηση που δόθηκε στη σχέση με την Κούβα και με, ξεκινώντας από την ε, ε αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και φτάνοντας και στην επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα του ειδικού εκπροσώπου. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι Μιλώντας ε, ο Ραούλ Κάστρο στα Ηνωμένα Έθνη την προηγούμενη εβδομάδα, ουσιαστικά έριξε το φταίξιμο σε κάθε ε, κογκρέσο γιατί ε, δεν αποκατέστησε τις σχέσεις και δεν ήρε το εμπάργο. Επομένως φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει ολοταχώς μια πορεία για την αποκατάσταση των σχέσεων. Και πρέπει να πω ότι ο Ομπάμα έκανε ότι, έχει, ε, έκανε παρά την αντίθεση των Ρεπουμπλικάνων και παρά το ε, πολύ ισχυρό λόμπι των, κατά της άρσης του εμπάργου. Ε, και εκεί έχουμε πολύ μεγάλη εκπροσώπηση και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία. Και πρέπει να πω ότι αυτό το παιχνίδι δεν είναι εύκολο, παρόλα αυτά τα κατάφεραν. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η Ευρώπη έχει ιστορικές σχέσεις με την Κούβα, συγκεκριμένες σχέσεις και δεσμεύσεις ενώπιον της Κούβας και κάποιες χώρες με την ιστορική κληρονομιά σχέσεών τους με την Κούβα, ουσιαστικά δείχνουν ότι είναι διατεθειμένες να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με την Κούβα. Και γι' αυτό ακριβώς ε, η Ευρώπη δεν θα έπρεπε να εκπλήσεται από άλλους θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματική και να είναι και λίγο πιο ρεαλίστρια στις σχέσεις της με την Κούβα και αντίστοιχα η Ευρώπη ε, συνειδητοποιεί απολύτως ότι σε καιρούς αλλαγής ε, και στη Λατινική Αμερική η Κούβα είναι ένας από τους μοχλούς πίεσες που διαθέτουμε προκειμένου να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στη Λατινική Αμερική γνωρίζοντας το ρόλο ε, είτε για καλό είτε για κακό που έχει διαδραματίσει η Κούβα εδώ και δεκαετίες. Γι' αυτό και κατά την άποψή μας θα πρέπει ε, να εξετάζουμε την Κούβα όχι μόνο βάσει συναισθημάτων ε, αλλά και με κάποιο αντίστοιχο βαθμό ρεαλισμού και να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο αποτελεσματικότητας ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή με θετικό τρόπο όχι μόνο για την Κούβα αλλά για τη Λατινική Αμερική. Και τρίτον, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι η Κούβα δεν είναι μόνη της και δεν ε, είναι αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ ΗΠΑ και ε, Ευρώπης. Η Κίνα είναι ε, πολύ σημαντική και έχει πολύ μεγάλη παρουσία αυτή τη στιγμή στη Λατινική Αμερική και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πολύ σύντομα θα έχει αντίστοιχη παρουσία και στην Κούβα, όπως επίσης και η Ρωσία. Εάν καθυστερήσουμε εμείς πάρα πολύ με τους προβληματισμούς μας, θα χάσουμε πάλι το παράθυρο ευκαιρίας για την ε, ε, δέσμευσή μας με την Κούβα και να κάνουμε αυτό το οποίο κάνουμε συνήθως με τη χώρα αυτή, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, εγώ είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι σε όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με και με θετικά, μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις στην Κούβα και θα έλεγα με ε, μεγάλο βαθμό φθόνου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε κατάφεραν να απελευθερέσουν ε, καταδίκους φυλακισμένους. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει να απελευθερήσουμε φυλακισμένους από τις φυλακές της Κούβας. Γιατί τα κατάφεραν αυτοί και εμείς από πλευρά Ευρώπης, είτε αποτύχαμε, είτε δεν είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Και τέλος, πρέπει να πω ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχητικές αλλαγές στη Λατινική Αμερική και με τη συνεργασία της Κούβας ίσως θα μπορούσαμε να τις διαχειριστούμε λίγο καλύτερα. Όπως για παράδειγμα την κατάσταση λόγω της τόσης οικονομίας στη Βραζιλία με τις περιφερειακές συνέπειες που έχει και το καθεξής. Η Κούβα είτε μας αρέσει είτε όχι, μόλις το είπατε κι εσείς και εγώ θα ήθελα και εγώ να το αναφέρω στην παρέμβασή μου, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματική ε, για την αντιμετώπιση της επιδημίας του έμπολα. Υπάρχουν αρκετοί γιατροί και εμπειρογνώμονες εκεί και ε, η αντιμετώπιση που έχουν αυτοί για την Αφρική διαφέρει και λίγο από την αντιμετώπιση που έχουμε εμείς και την οπτική, οπτικό πρίσμα το οποίο αντιμετωπίζουμε. Κατέφεραν λοιπόν να επηρεάσουν τα πράγματα και να συνεισφέρουν σε μια παγκόσμια κατάσταση. Ε, υπάρχει λοιπόν κοινό τόπος μεταξύ Ευρώπης και Κούβας και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και να έχουμε συνέχεια για το μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζούμπερ, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λέφλερ για την παρέμβαση του. εμείς έχουμε συναντηθεί και σε άλλα βήματα, ιδίως ε, στο πλαίσιο της Eurolab η ερώτηση θέλω να θέσω έχει δύο σκέλη. Καταρχήν, να πω ότι είναι προφανές ότι ζούμε σε μια ιστορική στιγμή επειδή εγκαταλείπονται μια σειρά πολιτικών απομόνωσης σε σχέση με τον κουβανικό, με τον κουβανικό λαό και θα πρέπει φυσικά να εγκαταλειφθούν αυτές οι πολιτικές γιατί έχουν αποτύχει. Και Επομένως, χρειάζεται μια αλλαγή της στρατηγικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Πολιτειών. Όμως, αν αυτό που θέλουμε είναι ένας εξομαλισμένος ε, διάλογος, τότε υπάρχουν εδώ δύο αχίλιες τέρνες. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τα δύο μέρη να μην μπουν έχοντας, επιδιώκοντας διαφορετικά πλεονεκτήματα. Άκουσα όλη τη διαδρομή που περιέγραψε ο κ. Λέφερ στις διαπραγματεύσεις με την Κούβα και είναι ουσιαστικά παράδοξο ε, το ότι δυσκολευόμαστε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις ε, με την ε, Κούβα. Ουσιαστικά μιλάμε εδώ για ένα πολιτικό εργαλείο που έχει μεγάλη συμβολική αξία και που διατηρείται όμως ουσιαστικά δεν έχει διπλωματική αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε ε, για τη δυνατότητα παρέκκλησης από αυτή την κοινή θέση και ποιες είναι οι δυνατότητες και προοπτικές να υπάρχει παρέκκληση από αυτή την κοινή θέση και αν ε, μπορεί να τεθεί στο Συμβούλιο αυτή η αναγκαιότητα από εσά και από την Κομισιόν. Τώρα η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το εμπάργκο. Το εμπάργκο δυστυχώς ακόμη παραμένει και στο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Κούβα, αλλά και με τι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος είναι ο ρόλο που έχει διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να τεθεί τέλο σε αυτό το εμπάργκο. Όπω είπε ο κ. Λεφλερ, αυτή είναι η πρόθεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί τέλο σε αυτό το εμπάργκο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, κ. Ζούμπερ. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε στον κύριο Λέφλερ το λόγο για να απαντήσει σε μία σειρά ε, ερωτήσεων, 10-12 λεπτά και μετά θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ομάδες. τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή πολιτική, το ρόλο της κοινή θέση, τις ε, ε, αλλαγές στις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών, τη σχέση μεταξύ των δύο, εξελίξεις ε, στο ίδιο το νησί και το συνολικό διεθνές πλαίσιο στο οποίο διαδραματίζονται όλα αυτά. Ο κύριος Γκάλερ είπε ότι ξαναδιάβασε την κοινή θέση και δεν ε, διαπίστωσε να υπάρχει κάτι ε, επίμαχο ε, εντός του κειμένου. Ναι, είναι ένα γενικό κείμενο το οποίο αναφέρει τις πάγιες ευρωπαϊκές θέσεις για την κοινωνία που θα θέλαμε να έχουν εταίροι μας. Δεν είναι κάποια δυσκολία, γιατί δεν λέει ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να κάνουμε κάτι, εκτός από το να προωθήσουμε κάποιο όραμα. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει κανείς ότι η αποτυχία της κοινή θέση είναι ότι συνήθως η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με τη δημοσίευσή της ε, στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα παράδοξο τρόπο, γι' αυτό και δεν έχουμε και τόσο πολλές κοινέ θέσεις. Αυτό το οποίο είναι σαφές, όταν μας έδωσε μια διαπραγματευτική εντολή το Συμβούλιο για τη Συμφωνία Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας, ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της προώθησης των αλλαγών και το να βοηθήσουμε να συνδράμουμε σε αυτές τις αλλαγές ε, στην Κούβα εξακολουθεί να ισχύει. Είναι αν θέλετε μια ε, εξαργύρωση όχι μιας ε, κοινή θέσης, μιας θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά το να προωθήσουμε τις αλλαγές είναι σημαντικό γιατί σημαίνει ότι ξεκινάει μια διαδικασία με τον εταίρο μας και ξεκινάει και μια διαδικασία όρων επί των οποίων θα ξεκινήσει ο διάλογος και περαιτέρω η συνεργασία. Πώς θα γίνει τώρα αυτό και τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Πολλοί από εσά θα γνωρίζετε ίσως ότι πριν από αρκετό καιρό τώρα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αλλά κάποιος Αμερικάνος δημοσιογράφος χαρακτήρισε την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ε, σαν ε, ήπια λόγια, ενώ ταυτόχρονα κρατά ένα τεράστιο καρότο κάποιος, ένα δώρο. Ε, εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί με τις τιμωρίες. Οι τιμωρίες ε, σπάνε και άμα δεν σπάνε τιμωρίες, σπάνε οι ίδιοι άνθρωποι και δεν μας αρέσει αυτό. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να μην φεύγουν και θέλουμε να κερδίσουμε τα επιχειρήματα μέσα της πυθούς και όχι ε, να τους υποχρεώνουμε να αλλάξουν. Εμείς δεν έχουμε τα μέσα να εφαρμόσουμε αλλαγές ε, πουθενά αλλού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να την προωθήσουμε, μπορούμε να την ενθαρρύνουμε την αλλαγή, αλλά στο τέλος Εάν μια χώρα, η κυβέρνησή της και ο λαός της, οποιαδήποτε χώρα και αν είναι αυτή, δεν δεσμευτεί, εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε για αυτούς. Αυτό ισχύει και για την Κούβα, αλλά ισχύει και για πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Και εδώ, ε, επιτρέψτε μου να πω ότι μάλλον υπάρχουν και αρκετές άλλες χώρες ε, στον κόσμο που Επίσης έχουν κυβερνήσεις ενός κόμματος από συγκεκριμένο ιδεολογικό παρελθόν ε, με τις οποίες έχει ξεκινήσει ακόμα και πρόσφατα συμφωνία συνεργασίας χωρίς καμία ένσταση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από Εθνικά Κοινοβούλια. Πρέπει να δεχτούμε ότι πράγματα συμβαίνουν ε, με διαφορετικές ταχύτητες ή πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας. Και βεβαίως αν ξεκινήσει πολιτικός διάλογος και υπάρξει συμφωνία συνεργασίας και πολιτικού διαλόγου, αυτό θα γίνει, όπως είπε και η κυρία Σακοράφα, μέσω μιας εταιρικής σχέσης. Το κατά πόσο θεωρείται ισότιμη η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 500 εκατομμυρίων και της Κούβας των 10 εκατομμυρίων είναι άλλη υπόθεση, αλλά σίγουρα θα είναι μια εταιρική σχέση σεβασμού. Σίγουρα. Βέβαια θα συμφωνείτε ότι ταυτόχρονα σε αυτή την εταιρική σχέση ε, και σε αυτό τον πολιτικό διάλογο εμείς θα υποστηρίζουμε τις θεμελιώδεις αξίες μας και οι θεμελιώδεις αξίες μας είναι το να μπορεί κάποιος να εκφράσει την άποψή του γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη και να προωθήσουμε αλλαγές σε μια κοινωνία. Θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τις αρχές αυτές στο διάλογό μας με την Κούβα και τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε συνεργασία με τις κουβανικές αρχές και με τους υπόλοιπους φορείς στην Κούβα. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε όσες περισσότερες πλευρές της κοινωνίας της Κούβας, αλλά ταυτόχρονα με σεβασμό στα πλαίσια του δικαίου. Δεν γίνονται πράγματα πίσω από την πλάτη του λαού και σίγουρα πίσω από την πλάτη του ίδιου του νόμου. Η προσέγγιση τώρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κούβας, όπως σας είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, είναι κάτι το οποίο είναι ευπρόσδεκτο. Είναι θετικό για την Κούβα, είναι θετικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θετικό για το ευρύτερο δυτικό ημουσφαίριο και είναι θετικό και για μας. Σε κάποιο βαθμό, κατά πάσα πιθανότητα, δυσκολεύει λίγο τις διαπραγματεύσεις μας, διότι οι εταίροι μας αποκτούν περισσότερη εμπιστοσύνη είναι πιο σίγουρη τώρα από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο. Και βεβαίω ε, τους ε, οθεί ε, και τους καταλαμβάνει αρκετό χρόνο η δυνατότητα συνεργασίας με τους εταίρους μας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στη Ναβάνα. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι σαφέ είναι ότι αυτό το οποίο συνέβη μεταξύ ΕΠΑ ε, και Κούβα ήταν η αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων. Όπω είπατε κι εσεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση ω Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διπλωματικέ σχέσει με την Κούβα εδώ και 30 χρόνια. Τα περισσότερα κράτη-μέλη για πολύ περισσότερο διάστημα. Εμεί βρισκόμαστε σε άλλο επίπεδο σχέσεων. αν βάλετε από τη μια μεριά το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, ε, με τον τρόπο που προχωράει βέβαια η Βενεζουέλα, κατά πάσα πιθανότητα θα το βάλει και η ίδια στο προσκήνιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, μακράν ο μεγαλύτερος εταίρος της ε, Κούβας, είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής της Κούβας, επομένως είναι ο πιο σημαντικός εταίρος για τις οικονομικές αλλαγές και τον οικονομικό εξυγχρονισμό. Και αυτό εξακολουθεί να ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει για αρκετό καιρό. Επίσης είναι σαφές ότι καθώς η, Κίνα, η Κούβα προωθεί στενότερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναλύει και τις προοπτικές για το πώς μπορούν να διαμορφωθούν οι σχέσεις πέραν του εμπάργου, θα αντιληφθούν σίγουρα σαφώς ότι στην ιστορία του 20ου αιώνα τα πρώτα 50 χρόνια εξαρτώνταν πλήρως από αυτό το μεγάλο βόρειο εταίρο και το δεύτερο ήμιση του αιώνα εξαρτώνταν από μια άλλη μεγάλη χώρα λίγο μακρύτερα. Και οι δύο αυτές εξαρτήσεις αποτέλεσαν αποτυχία για την Κούβα με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά αυτό το αντιλαμβάνονται πλήρως και αντιλαμβάνονται ότι την επόμενη φορά δεν θα πρέπει να εναποθέσουν όλες τις ελπίδες τους σε έναν και νομίζω ότι αυτό θα ενισχύσει και τα συμφέροντά τους για συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να το αποδυναμώσει. Διότι θεωρούν ότι εμείς είμαστε ένας χρήσιμος επιπλέον εταίρος και μάλιστα κάποιος ο οποίος τους είναι οικείος και κάποιος ε, τον οποίον εμπιστεύονται σε γενικές γραμμές. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε ότι θα χάσει το ενδιαφέρον της η Κούβα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα απομακρυνθεί όχι λόγω των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι λόγω της Ρωσίας, η οποία ε, πόρο απέχει από το να αποκαταστήσει τις σχέσεις που είχε πριν από 20 χρόνια με την Κούβα ή και την ίδια την Κίνα. Εμείς χαιρόμαστε για την περαιτέρω και ισχυρότερη εμπλοκή της Κίνας ως επενδυτικό εταίρο, ως οικονομικό εταίρο, ακόμα και ως ε, εταίρο συνεργασίας θεωρούμε ότι αυτά είναι θετικά νέα. Αλλά σίγουρα υπάρχει πολύ περισσότερος χώρος για όλους μας. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ανησυχούμε για το θέμα αυτό. Τώρα, η διπλή αυτή μετάβαση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ντεσαρνές, οικονομική και δημοκρατική μετάβαση. Απόλυτα ορθό και νομίζω ότι είναι αλληλένδετα τα δύο και δεν θα υπάρξει επιτυχία του ενός χωρίς το άλλο εν τέλει. Δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πλήρω τον εξυγχρονισμό ε, χωρίς ε, την υποστήριξη του ενός από το άλλο και νομίζω ότι αυτό δεν το πιστεύουν ούτε οι ίδιες οι αρχές της Κούβας και νομίζω ότι εδώ έρχεται και το στοιχείο της συνέχειας. Μπορεί να εξυγχρονιστεί το παρόν σύστημα και να γίνει πιο αποτελεσματικό, πιο δυναμικό, να δημιουργεί θέσεις εργασίας και να γίνει ανταγωνιστικό διεθνώς, χωρίς να αλλάξει η ουσία οικονομική και η γεωπολιτική. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα ανά τον κόσμο που θα τους καθησυχάσουν αν μένουν σε αυτή την άποψη, τουλάχιστον όπως το, το βλέπουμε εμείς το ζήτημα. Μπορεί βέβαια εμείς ε, να περιοριζόμαστε στην προοπτική μας από την προσωπική μας εμπειρία. Εμείς προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε νέο σκεπτικό, νέους τρόπους εργασίας, για παράδειγμα στα προγράμματα σε θέματα γεωργίας, ε, σε συνεργασία με συνεταιρισμούς ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι συνεταιρισμοί θα λαμβάνουν περισσότερο περιθώριο για ανεξάρτητες κινήσεις ώστε να μπορούν να αποφασίζουν σε τοπικό επίπεδο και να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι όχι μόνο για την παραγωγή αλλά και για την πώληση των προϊόντων τους. Ε, αλλά αυτό ε, είναι κάτι το οποίο θα καθυστερήσει πάρα πολύ να υλοποιηθεί. Πόρο απέχουμε. Και ε, εξίσου μακρινή είναι η διαδικασία και σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν αλλαγές εν εξελίξη, υπάρχει πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και κάποιων αντιπροσωπευτικών δομών που σίγουρα δεν θα ολοκληρωθούν βραχυπρόθεσμα δεν θα έχουμε δομές οι οποίες ε, θα μοιάζουν αυτή τη στιγμή με αυτές που γνωρίζουμε. Σίγουρα όμως αποτελεί ευκαιρία και αποτελεί ευκαιρία για δημόσια συζήτηση για το προς τα που θέλουν να κατευθυνθούν. Και θεωρώ ότι για μας ένα από τα πιο ουσιαστικά ζητήματα είναι να κάνουμε όσες προσπάθειες μπορούμε προκειμένου να διευρύνουμε το χώρο για δημόσια συζήτηση προς το συμφέρον των κουβανών και της κοινωνίας ε, της Κούβας εν γέννη. Να γίνει περισσότερη συζήτηση λοιπόν για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας, το οποίο θα μας επιτρέψει εμάς να βρούμε νέους τρόπους να τους βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό θα γίνει και στο πολιτικό πλαίσιο αλλά και στο οικονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Μιλανμόν Μον αναφέρθηκε στον οικονομικό πυλώνα. Όπως σας είπα, δεν πρόκειται για προτιμησιακή συμφωνία, γιατί δεν μας ζητήθηκε και ποτέ τέτοια συμφωνία. Και σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο με την κατάσταση της ε, οικονομίας αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε πώς θα εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επενδυτές θα μπορούν να επενδύσουν με παραγωγικό τρόπο και γνωρίζοντας ότι δεν θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού πολύ γρήγορα. Υπήρξε ένας νέος επενδυτικός νόμος στην Κούβα πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο και κάτι. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη κατεύθυνση, αλλά σίγουρα πρέπει να αποκτήσει και ισχυρότερες δομές. Υπάρχει επίσης η διευκόλυνση του εμπορίου. Η βοήθεια προς τους κουβανούς οικονομικούς φορείς ε, και τους νέους ανεξάρτητους ή μη ανεξάρτητους φορείς να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους δίνονται στην Ευρώπη με καλύτερο τρόπο από ό,τι μπορούσαν μέχρι τώρα να αντιληφθούν πώς ε, λειτουργούν οι ευρωπαϊκές αγορές, ε, τα ευρωπαϊκά μοντέλα κατανάλωσης ώστε να υπάρχει ε, μια βελτίωση και μια συνέχεια ώστε να μπορέσουν να ικανοποιήσουν και τις προσδοκίες των ευρωπαϊκών αγορών. Πρόκειται για τομείς οι οποίοι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν πολύ, πρόκειται για τομείς ε, στους οποίους ε, μπορούμε να δημιουργήσουμε και γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ της κουβανικής διοίκησης ε, από το τεχνικό επίπεδο ε, σταδιακά στο επίπεδο χάραξης πολιτικής. Κάτι το οποίο θα έρθει να προσθεθεί και στο διάλογο για τις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και τις περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές ε, στην οικονομία της Κούβας και στην κοινωνία της Κούβας. Θα καθυστερήσει αυτό, αλλά εμείς έχουμε υπομονή και θα τους βοηθήσουμε σύν το χρόνο ε, περαιτέρω ε, εξυγχρονιστικά μέτρα στην Κούβα προς το συμφέρον των Κουβανών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λέφλερ, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις συνεισφορές σας. Νομίζω ότι ήταν ε, πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση για τις εξελισσόμενες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας και δεδομένου ότι και μόλις υλοποιήθηκε και ο πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων ε, πριν ένα μήνα στην Κούβα. Στην αποστολή στην οποία ήσασταν επικεφαλής κύριε Λεφλερ επίσης, ε, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα για τη Λατινική Αμερική και τη συνεργασία με την Λατινική Αμερική και κάτι που ενθαρρύνεται και από τον προϋπολογισμό και αν ε, μια μέρα έχουμε σεβασμό των δικαιωμάτων και ελεύθερες εκλογές στην Κούβα, νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ θετικό και θα έχουμε συνεισφέρει σε αυτό. Λοιπόν, αύριο θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας στις 9 και θα περάσουμε και στην ψηφοφορία για το ρόλο της έντασης των Ηνωμένων Εθνών στις 10